Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Εάν δεν έχετε αντίρρηση. Χρειαζόμαστε όμως λίγο χρόνο. Πρέπει να ετοιμάσουμε ένα έγγραφο επί τη βάση της απόφασης των συντονιστών Στα σημεία 1 και 2 δεν έχουμε τίποτα. Και το 3 μπορούμε να το εγκρίνουμε, οπότε να εντάξει η ημερησία διάταξη. 23 Ιανουαρίου, 22 και 23 Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου επίσης είναι τα πρακτικά. Μπορούμε να εγκρίνουμε αυτά τα πρακτικά. Σημείο 5. Ανακοινώση του Προέδρου. Τίποτα δεν έχω να σας ανακοινώσω. Πληροφορίες για τις αποφάσεις των συντονιστών. Και εδώ θέλω να σας πω ορισμένα πράγματα. Πρωτού ψηφίσουμε, θα πρέπει να, να μια επιστολή που συμφωνήθηκε στη συνάντηση των ε, συντονιστών, αλλά δεν έχει διανεμηθεί από ό,τι γνωρίζω. Και θα ψηφίσουμε μετά για τα τρία πιλωτικά προγράμματα, τα οποία είναι μέσα στα έγγραφα που έχουμε Α, υπάρχει μια νέα μορφή. Η πρόταση του ΕΛΚ έχει γίνει δεκτή. Και η παράγραφος 9 επίσης ανακρίθηκε στις συνεδρίες των συντονιστών. Και τώρα μία ακόμα ανακοίνωση. Πήραμε μια απόφαση ως συντονιστές. Επειδή είναι η τελευταία μας συνεδρίαση της Επιτροπής μας και η τελευταία φυσικά συνεδρίαση των συντονιστών, αν χρειάζεται να, κάνουμε κάποια, να πάρουμε κάποια απόφαση, θα την πάρουμε με γραπτή διαδικασία αν υπάρχει κάτι πάρα πολύ κατεπήγον, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μια συνεδρίαση έκτακτη, αλλά προς το παρόν δεν προβλέπουμε να χρειαστεί να κάνουμε κάτι τέτοιο, προτού συγκροτηθεί η νέα μας Επιτροπή. Αλλά νομίζω ότι προς το παρόν η γραφή διαδικασία είναι εντάξει. Σημείο 6 τώρα. Θα το πω στα αγγλικά. Υπήρχε αυτή η επιστολή που ζητούσε από την πλευρά του ΕΛΚ να τροποποιηθεί παράγραφος 7 ενεκρίθη στη συνεδρία των συντονιστών με πλειοψηφία και στην παράγραφο 9 Είχε εγκριθεί και εκεί με μια πλειοψηφία στη συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε αυτή είναι η επίσημη πρόταση των συντονιστών. Αλλά επειδή δεν το έχετε δει το έγγραφο αυτό, χρειάζεται δύο-τρία λεπτά για να το διαβάσετε. Εντάξει. φαίνεται λίγο παράξενο. Τώρα νομίζω ότι έχετε την τελευταία, την πιο πρόσφατη εκδοχή. Είναι λοιπόν μια επιστολή που έχουμε βάλει στο σύστημα. Βλέπετε λοιπόν τη νέα πρόταση. Κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απλώς θα σας πω ότι η πολιτική μου ομάδα, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, θα υπερψηφίσει αυτή την επιστολή, αλλά είναι εναντίον της 7ης παραγράφου σε αυτή την επιστολή, δηλαδή για την ε, αλλαγή αυτή που έχει εισαχθεί στην 7η παράγραφο. Ευχαριστώ. Yes, I will, because during... Εντάξει. Είχε σταλεί σε όλους τους συντονιστές και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας το ΕΛ και οι σοσιαλιστές πρότειναν δύο αλλαγές, μία στην παράγραφο 7 και η άλλη στην παράγραφο 9. και εγώ αν θέλει κάποιος να προτείνει κάτι σχετικό θα το αντιμετωπίσω σαν τροπολογία σε αυτή την πρόταση και μετά πρέπει να ψηφίσουμε την παράγραφο την πρόταση του ΕΛΚ για την παράγραφο 7. Να δούμε αν δεχόμαστε την τωρινή πρόταση των συντονιστών ή την προηγούμενη. Αλλά λέω η πρόταση του ΕΛ και των σοσιαλιστών ώστε να ξέρουν όλοι περί πρόκειται. Επισήμως στη συνάντηση των συντονιστών είπαμε επί τη βάση της πρότασης των συντονιστών του ΕΛΚ, συγγνώμη. Οπότε έχουμε μια πρόταση του ΕΛΚ και μια πρόταση των σοσιαλιστών. Κυρία Κονέλσε, θέλετε να πείτε κάτι. Να σας πω απλώς ότι είχαμε κάποια συζήτηση για τη λέξη ε, segmentation έναντι της λέξης segregation, δηλαδή κατάτμιση και όχι ε, διάκριση. Η segmentation, κατάτμιση σημαίνει κάτι διαφορετικό από την ε, segregation, δηλαδή την, ε, τον διαχωρισμό. Είναι λοιπόν τελείως διαφορετική έννοια. Αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε σε αυτήν την παράγραφο είναι περισσότερο ο διαχωρισμός σε διαφορετικές ομάδες εργασιών και όχι κατάτμιση σε διάφορα επίπεδα. Θα υποστήριζα λοιπόν την αρχική μορφή και όχι τη μορφή του ΕΛΚ. Αλλά τουλάχιστον να ξαναγυρίσουμε στη λέξη segregation, διαχωρισμό σε αυτήν την περίπτωση. Είναι προφορική τροποποίηση αυτό. Ναι. Ζητώ να γίνει αυτή η αλλαγή, το segregation, το segmentation να γίνει segregation. νομίζω ότι θα μπορούσα να προτείνω μια συμβιβαστική λύση. Αν έχουμε και segmentation και segregation, για να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι για τα θέματα αυτά. Δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτή τη συζήτηση και δεν θέλω να υπάρξει συζήτηση για το θέμα αυτό. ήταν σαφές στη συνάντηση των συντονιστών ότι συζητήσαμε για το θέμα του segmentation και segregation και ήταν διαφορετικές οι απόψεις οι οποίες διατυπώθηκαν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να, να καταλήξουμε τώρα σε μία λύση. Αν δεν θέλετε τη μία λέξη θα την ακυρώσετε και αν δεν θέλετε την άλλη λέξη και αυτή μπορείτε να την ακυρώσετε. Κύριε Χάνιμπολ. Σχολαστικό είναι αυτό που λέω αλλά η λέξη segmentation δεν είναι αγγλική λέξη, εν πάση Μήπως μπορούμε να πούμε σπάσιμο στα δύο, διαχωρισμός. Ή σας δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό. Εγώ θα τη δω την πρόταση της κυρίας Κονέλση σαν προφορική τροπολογία και μετά ψηφίσουμε. Οπότε αν θέλετε την segmentation έχετε segmentation, αν θέλετε segregation έχετε segregation. Ζούμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μου θα υποστηρίξει την πρόταση αυτή, δηλαδή να έχουμε την ε, segregation στη θέση του segmentation. Η έρευνα η οποία έγινε για τις συνθήκες εργασίας αναφέρει στο σημείο 1 την διάκριση βάση φύλου. Αυτή λοιπόν πρέπει να είναι η διατύπωση που θα χρησιμοποιήσουμε. Και δεν νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όπως ε, θέλησαν ορισμένα να δημιουργήσουν την εντύπωση στη συνεδρίαση των συντονιστών. Θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε το αρχικό κείμενο στην παράγραφο 7 Το αρχικό κείμενο λοιπόν που λέει υπογραμμίζει ότι η κατάλληλη χρηματοδότηση θα πρέπει να προβλέπεται για ενέργειες οι οποίες έχουν σαν στόχο να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις της κρίσης. Ελπίζω ότι όλα είναι σαφή. και θα το αντιμετωπίσω λοιπόν αυτό σαν ένα σύνολο από παραγράφους πρέπει να ψηφίσουμε τη μία μετά την άλλη. Ελπίζω ότι δεν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις για αυτές τις παραγράφους από την 1 ως την 6. Μπορούμε να ψηφίσουμε αυτές από κοινού, την 1 ως 6. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα η επίμαχη παράγραφος 7. Πρώτα απ' όλα, προφορική τροπολογία και μετά η πρόταση του ΕΛΚ εναντίον της πρότασης των σοσιαλιστών. Και αν κερδίσει η πρόταση του ΕΛΚ, τότε εκπίπτει η πρόταση των σοσιαλιστών. Και θα περάσουμε στις παραγράφους 8 και 9. Η πρόταση του, των σοσιαλιστών είναι το αρχικό κείμενο και του ΕΛΚ το τροποποιημένο κείμενο όπως έχει εγκριθεί από τους συντονιστές πριν από 20 λεπτά. Θέλετε να πείτε κάτι. Εξ ονόματος του ΕΛΚ θέλω να πω ότι πρέπει να ψηφίσουμε χωριστά και την Ενέα. Εντάξει. Κάτι δεν είναι πολύ σαφές. Τι ψηφίζουμε τώρα όλη την παράγραφο ή μόνο την προφορική τροποποίηση. Πρώτα την προφορική τροποποίηση. Και μετά θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το segregation εναντίον του segmentation. Αυτό είναι ένα κείμενο που δεν μπορέσατε να δείτε προηγουμένως. Γι' αυτό σας αφήνω να καταθέσετε προφορικές τροπολογίες. Δεν θα είμαι ευτυχισμένο αν έχουμε τόσες πολλές τροπολογίες όμως. Φυσικά έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε προφορικές τροπολογίες. Και οτιδήποτε είναι διαφορετικό από το αρχικό κείμενο, το αντιμετωπίζω ως τροπολογία. Μπορεί όλα αυτά να μην είναι πολύ σαφή. Πρώτα την προφορική τροπολογία και μετά το σύνολο της παραγράφου. Και αυτό θα εξαρτεί από το αν εγκριθεί η τροπολογία ή όχι. Είναι σαφές. Αν υποστηρίζετε για την διατύπωση segregation, διαχωρισμός, πρέπει να πείτε ναι σε αυτή την τροπολογία. Αν θέλετε το segmentation κατάτμιση να πείτε όχι. Εντάξει. Ποιοι είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Κατά. Αν θέλετε τη λέξη segregation, λέτε ναι. Segmentation πρέπει να πείτε όχι. υπέρ και πάλι. Κατά. Η πλειοψηφία υποστηρίζει το segregation, διαχωρισμός. Εντάξει. Τώρα ψηφίσουμε όλη την παράγραφο με τη λέξη segregation. Δεν υπάρχει segmentation, ψηφίζουμε με segregation. Μόνο το ΕΛΚ ψήφισε υπέρ του segmentation. Μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο αν επιμένετε. υπέρ του segregation. Κατά του segregation για segmentation δηλαδή. Μάλιστα. Οπότε κερδίζει η, δια, η διατύπωση διαχωρισμός, segregation. Ψηφίζουμε τώρα την παράγραφο 7. Και για να το κάνω σαφέ, Έχουμε την πρόταση του ΕΛΚ. Η πρόταση του ΕΛΚ είναι η πρόταση των συντονιστών. Και βγάζουμε αυτό ότι λαμβάνουμε υπόψη τα αποτελέσματα της κρίσης και βάζουμε το ε, καινοτόμοι τομεί όπως ο τομής της πληροφορικής. Ποιοι είναι υπέρ τη πρόταση του ΕΛΚ. Κατά. Πρέπει να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Θα προσθέσω τη δική μου ψήφο γιατί δεν έχω κάρτα μαζί μου. Πέρα τη ψηφοφορία. Η ισοψηφία άρα απορρίπτεται. 7-7. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την πρόταση των σοσιαλιστών. Υπέρ της πρότασης των σοσιαλιστών, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος άρχεται ηλεκτρονικά. Πέρας. Και εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Και πάμε στην επόμενη ψηφοφορία για τα πιλωτικά προγράμματα. Έχουμε τρία πιλωτικά προγράμματα. Ζήτησα να τα πάρουμε συνολικά. Όχι, δεν γίνεται. Ένα προς ένα. Αυτό που πρότεινε η Τσίτα Γκουρμάη. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρόταση Κορνέλισεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και το τρίτο υπέρ κατά. Εδώ είναι ασαφές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελειώσαν οι ψηφοφορίες. Βγαίνουμε στο σημείο υπαριθμών 8. Okay, then we, then Σημείο υπαριθμών 8 και χαιρετίζω την κυρία Μανουέλα Σακ από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας στην Ιταλία. Προσπάθησα να το πω και ιταλικά, αλλά αστόχησα. Θα μας παρουσιάσετε τη μελέτη για το mainstreaming, την εισαγωγή της διάστασης του φύλου στις επιτροπές και αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να παρουσιάσουμε τη μελέτη μας. Εγώ και η Φλάβια Πέσε αναλάβαμε αυτήν την μελέτη μαζί με τον επιστημονικό σύμβολο Μπρούνο Βέντε. Θα προσπαθήσω να σας το παρουσιάσω σύντομα γιατί η μελέτη είναι περίπλοκη, αρκετά περίπλοκη. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό η Επιτροπή των γυναικών συνέβαλε στην εφαρμογή του mainstreaming του φύλου στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ανάμεσα δηλαδή τον Ιούλιο του 2011 και τον Ιούλιο του 2013. Θεωρήσαμε ε, εξετάσαμε λοιπόν αυτό που μας ε, ζητήθηκε. Χρησιμοποίησαμε την προσέγγιση της ανάλυσης πολιτικής και για να διεξάγουμε αυτή τη μελέτη, ε, μελετήσαμε τη συγγετική τεκμηρίωση και αυτό ήταν αρκετά δύσκολο να καταλάβουμε πώς και ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθείτε εδώ ώστε να λάβετε αποφάσεις. Επίσης, εξετάσαμε τις νομοθετικές και μη νομοθετικές πράξεις που, ε, που καταρτίζει η Επιτροπή ΦΑΜ και τις, οι άλλες πέντε επιτροπές που μας υποδείχθηκαν στην, ε, κατά τον διαγωνισμό. Ε, εξετάσαμε στοιχεία, την ε, σύσταση των επιτροπών, ε, των αντιπροσωπείων από το διαδίκτυο και από τα site του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάναμε και κάποιες μελέτες, μάλλον συνεντεύξεις με συγχωρείτε, με ευρωβουλευτές αλλά και εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και επισκεφθήκαμε τα γραφεία του Κοινοβουλίου στις διάφορες χώρες για να δούμε πώς ε, αναπτύσσονται και πώς προτείνονται τα θέματα ε, ε, του φύλου και πώς προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πώς προβάλλονται. what the, our understanding of what... Τι καταλάβαμε λοιπόν για το πώς γίνεται το gender mainstreaming στο Κοινοβούλιο και ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής των Γυναικών. Το βασικό μας συμπέρασμα είναι ότι μπορούμε να δούμε ένα αρκετά ανεπτυγμένο νομικό σύστημα που στηρίζει το mainstreaming του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο όσον αφορά τα ίδια τα σώματα που ασχολούνται με το θέμα, αλλά και όσον αφορά, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένε επιτροπέ ομάδε που στηρίζουν το mainstream εντό του κοινοβουλίου, ωστόσο υπάρχει χώρο για βελτίωση. Έχουμε ένα πλαίσιο λοιπόν, το οποίο είναι πολύ καλά δομημένο, αλλά μπορεί να υπάρξουν ακόμα κάποιε βελτιώσει. Υπάρχει η Επιτροπή λοιπόν των Γυναικών που είναι το κεντρικό όργανο επιφορτισμένο με την προώθηση του mainstreaming στην νομοθετική και μη νομοθετική διαδικασία του Κοινοβουλίου. Υπάρχει η ομάδα υψηλού για την ισότητα των φύλων και την, και την ε, ε, διαφορά που συμπληρώνει κατά κάποιο τρόπο τις εργασίες της Επιτροπής Γυναικών γιατί εφαρμόζει το mainstreaming στις ίδιες τις δομές του Ευρωκοινοβουλίου και δεν έχει ρόλο να παίξει στο νομοθετικό, στην νομοθετική διαδικασία και μετά υπάρχει το δίκτυο του mainstreaming όπου συμμετέχουν πρόεδροι, αντιπρόεδροι κάθε μόνιμης επιτροπής και επηρεάζει την εργασία των άλλων επιτροπών και των υπολείπων διοικητικών σωμάτων. Αυτά τα τρία σώματα λοιπόν είναι σημαντικά. για το mainstreaming στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν εξετάσει κανείς το ρόλο της Επιτροπής Γυναικών και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο Κοινοβούλιο για την εφαρμογή του mainstreaming, υπάρχουν τρεις βασικές κρίσιμες πτυχές που προκύπτουν και που θα πρέπει να εξεταστούν. Τις λάβαμε λοιπόν αυτές υπόψη, τα βαλάβαμε υπόψη αυτά τα κεντρικά θέματα στις συστάσεις που προτείνουμε στο τέλος. Η πρώτη είναι ο ρόλος της Επιτροπής ΦΑΜ την διαδικασία σχηματισμού πολιτικής. Και εδώ υπάρχει ένα παζάρι στην ουσία, γιατί η Επιτροπή των Γυναικών έχει μια παράξενη οριζόντια ε, θέση, έχει αρμοδιότητες για τα δικαιώματα των γυναικών και για την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς της πολιτικής και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το mainstreaming. Ωστόσο, σπανίως είναι αρμόδια για νομοθετικές διαδικασίες, γιατί λίγες είναι οι νομοθεσίες που άμεσα αφορούν την ισότητα. Η βασική της δραστηριότητα εστιάζεται στο να επηρεάσει τις εργασίες άλλων επιτροπών μέσω γνωμοδοτήσεων ή τροπολογιών που στόχο έχουν το mainstreaming των ε, ε, φύλων. Αυτό σημαίνει πως η βασική δραστηριότητα της Επιτροπής ε, ε, ΦΑΜ είναι να προσπαθήσει να πείσει τις άλλες ε, επιτροπές να λάβουν υπόψη τους το θέμα της ισότητας των φύλων και του φίλου γενικότερα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η προσπάθεια που γίνεται να επηρεάσει την νομοθετική διαδικασία. Βέβαια, οι γυναίκες που είναι μέλη της Επιτροπής Γυναικών, ή μάλλον οι ευρωβουλευτές που είναι μέλη της Επιτροπής Γυναικών, είναι ταυτόχρονα μέλη και άλλων επιτροπών και έχουν δυνατότητα να προωθούν τις ε, γνωμοδοτήσεις αλλά και τις τροπολογίες για το mainstreaming στις άλλες επιτροπές. Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ βαρύς ο φόρτος εργασίας για τα μέλη αυτής της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει πως τα μέλη αυτής της Επιτροπής πρέπει να είναι πάρα πολύ ε, προσιλωμένα στα θέματα του, της ισότητας για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και από την ανάλυση που κάναμε. Αυτή η δέσμευση και αυτή η αφοσίωση υπάρχει. Δηλαδή πραγματικά η, τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών είναι αφοσιωμένα στο έργο τους, στην εργασία τους. Εξετάζοντας τώρα τον ε, ρόλο των Ευρωβουλευτών στην Επιτροπή των Γυναικών όσον αφορά το σχηματισμό πολιτικής ε, και στις διαδικασίες της νομοθετικής και της μη νομοθετικής του Κοινοβουλίου υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν και είναι πολύ σημαντικά διότι επηρεάζουν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής των Γυναικών στην προώθηση του mainstreaming. Πρώτη σημαντική φάση είναι η αρχική φάση, όπου οι διαδικασίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η διάσκεψη των Προέδρων επιλέγουν την αρμόδια επί τη ουσία επιτροπή και την γνωμοδοτική επιτροπή για κάποιο συγκεκριμένη πράξη, νομοθετική πράξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε αυτή τη φάση, μπορεί να υπάρξει και κάποια απόφαση Μάλλον, να υπάρξει περίπτωση όπου δύο επιτροπές ασχολούνται με την πρόθεση συγκεκριμένου νομοθετήματος. Αυτή η αρχική φάση είναι πολύ σημαντική, διότι σημαίνει ότι εκεί όπου η αποφασίζεται αν και κατά πόσο η Επιτροπή των Γυναικών πρέπει απλά να χρωμοδοτήσει ή αν θα επηρεάσει με υποβολή τροπολογιών κτλ. Η Επιτροπή των Γυναικών κατά την περίοδο που εμείς αναλύσαμε ως αρμόδια από τη Ουσίας Επιτροπή ε, ασχολήθηκε μόνο με τέσσερις ε, ε, εκθέσεις διαπιστώσαμε ότι η αποτελεσματικότητα των γυναικών, της Επιτροπής Γυναικών για την Προώθηση του mainstream των φίλων είναι μεγαλύτερη εκεί όπου ενεργεί ως συναρμόδια επιτροπή. Για να υποστηριχτεί λοιπόν η, η, να υποστηριχτεί ο ρόλος της Επιτροπής των Γυναικών θα πρέπει η Επιτροπή των Γυναικών να ε, ε, ορίζεται περισσότερο ως συναρμόδια επιτροπή. Επίσης, η γραμματεία της Επιτροπής έχει σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτή την αρχική φάση. και όπου δηλαδή λαμβάνεται η απόφαση στην διάσκεψη των Προέδρων. Είναι μια πολύ σημαντική φάση λοιπόν και υπάρχουν εδώ ξεκάθαροι ρόλοι που θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Δεύτερη ουσιώδης φάση είναι η ταύτιση, ο ορισμός των εισηγητών που αναλαμβάνουν γνωμοδοτήσεις ή εκθέσεις. Και εδώ η αξιοπιστία και η σημασία των εισηγητών της Επιτροπής ΓΙΝ είναι ιδιαίτερα σημαντική για θέματα βέβαια ισότητας των φύλων. Η επιλογή λοιπόν ενός καλού εισηγητή για τα διάφορα θέματα που πρέπει να αναλυθούν είναι πολύ σημαντική πτυχή της δουλειάς τους ένας επιτυχής εισηγητής τουλάχιστον από τις περιπτώσεις που αναλύσαμε είναι ένας ευρωβουλευτής που έχει σωστή και επαρκή γνώση τη δυνατότητα δικτύωσης ιδίως σε άτυπες συνθήκες, να έχει καλές σχέσεις δηλαδή με συναδέλφους του σε όλες τις επιτροπές όχι μόνο στη δική του πολιτική ομάδα αλλά και στις άλλες. Δικτύωση λοιπόν πολύ σημαντικό, πολιτικό πρεστίζ και αφοσίωση στην ιδέα της ισότητας των φίλων. Οι περιπτώσεις που θεωρήσαμε επιτυχής ως παρεμβάσεις οφείλονταν στη δυνατότητα του εισηγητή ή της εισηγήτριας να εφαρμόσει όλες αυτές τις αρετές. Άλλοι παράγοντες σε αυτή τη φάση είναι οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων, διότι εκείνοι αποφασίζουν πώς θα κατανεμηθούν οι εκθέσεις στα μέλη με το σύστημα των πόντων που είναι πολύ πολύπλοκο βέβαια και η γραμματεία επίσης που χορηγεί, προμηθεύει την τεχνική βοήθεια. Αυτές οι δύο φάσεις είναι οι σημαντικότερες για την αποτελεσματικότερη δράση της Επιτροπής ΓΙΝ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και ένας ακόμη παράγοντας λίγο εκτός του ρόλου των Επιτροπής ΓΙΝ, είναι πώς ακούγονται όλα αυτά στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης. Είδαμε ότι συνήθως όταν τα θέματα ισότητας των γυναικών συζητιούνται ήδη δημόσια και στα μέσα, τότε είναι πιο εύκολο για τις γυν να είναι αποτελεσματικές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όπως το να τους ζητηθεί να συμμετάσχουν σε κάποια μεικτή επιτροπή ή κάποια γνωμοδοτική επιτροπή. Βέβαια, αυτό είναι εκτός των αυστηρών δικαιοδοσιών των γιν, αλλά μπορούν και αυτές να κάνουν κάτι για να ακουστεί η άποψή τους για το θέμα της ισότητας των φύλων. Ο ρόλος λοιπόν της Επιτροπής γίνει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων η σημασία των εισηγητών και η ορατότητα της συζήτησης στο κοινό. Αυτά είναι οι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της δράσης των γυναικών για την ισότητα. Μετά εξετάσαμε τι έγινε από την Επιτροπή Γιν στην περίοδο που αναλύσαμε, Ιούλιο 2011 με Φεβρουάριο 2013. Και βλέπουμε ότι εξετάσαμε γνωμοδοτήσεις, τροπολογίες, εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας και μεικτή κοινή κοινοβουλευτική δράση. Οι γνωμοδοτήσεις είναι η κύρια δραστηριότητα κατά την περίοδο αυτή. 33 γνωμοδοτήσεις συμπληρώθηκαν. Και διατέθηκαν στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. 40 γνωμοδοτήσεις διεκπαιρεώθηκαν, αλλά μόνο 33 συμπληρώθηκαν. Αναλύσαμε λοιπόν τις 33 αυτές γνωμοδοτήσεις. Αυτές σχετίζονταν με 11 επιτροπές, γνωμοδοτούσαν προς 11 άλλες επιτροπές και πάνω από 700 τροπολογίες κατατέθηκαν για αυτές. Βλέπετε από τους αριθμούς αυτούς ότι προσπαθήσαμε να ταξινομήσουμε τα θέματα που εθίγησαν στις τροπολογίες και το κυριότερο ήταν τα δεδομένα και τα εργαλεία για τα φύλλα. Δηλαδή όλα τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τονιστεί το θέμα της ισότητος των φύλων, στατιστικά, στοιχεία, συστήματα εποπτείας, αξιολογήσεις, μεθοδολογίες κλπ. Και αυτά αντιπροσώπησαν παραπάνω από 50% των προτάσεων και τροπολογιών. Το άλλο μισό αφορούσε οικονομική και κοινωνική συμπερίληψη των γυναικών. Βλέπετε ότι τα υπόλοιπα θέματα ήταν πολύ λιγότερο σημαντικά στις τροπολογίες όπως οι υπηρεσίες, οι θέματα παιδείας και εκπαίδευση, ανθρώπινα δικαιώματα. Και κυρίως η βία κατά των γυναικών. Σε ορισμένε περιπτώσει, όπω είναι η περίπτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το γεγονό ότι υπάρχει μια άλλη επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι η επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αυτό εξηγεί γιατί δεν υπήρξαν τόσε πολλέ τροπολογίε και προτάσει που εκπορεύθηκαν από την Επιτροπή Γυναικών. Και εδώ μπορείτε να δείτε, αν μπορείτε να δείτε, ποιες επιτροπές ήταν αυτές που δέχτηκαν τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Γυναικών και πόσες τροπολογίες ενεκρίθησαν εν μέρη ή πλήρως και γενικά βλέπετε ότι περίπου ένα τρίτο, δηλαδή 29% ενεκρίθησαν. Δεν είναι τόσες πολλές. Γι' αυτό λέμε ότι μπορούν να υπάρχουν χώρος για βελτίωση. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην έγκριση των γνωμοδοτήσεών σα που καταδαπανούν πολύ χρόνο, απαιτούν πολύ εργασία. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι περισσότερε από αυτέ τι προτάσεις την χάνουν έγκρισης. Όπως βλέπετε η Επιτροπή Απασχόλησης, ΕΜΠΛ, ήταν αυτή η οποία ε, αντιμετώπισε τις περισσότερες προτάσεις και γνωμοδοτήσεις αλλά οι επιτροπές όπου υπήρξε το μεγαλύτερο ποσοστό ένκρισης είναι η Επιτροπή, Ελέγχου του Προϋπολογισμού και η Νομική Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν κάποιες στατιστικές που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Και στο τελευταίο, στην τελευταία στήλη Έχουμε τον αριθμό γυναικών σε κάθε επιτροπή για να δούμε αν υπάρχει μια σχέση, μια συσχετισμό ε, μεταξύ της ισορροπίας των φύλων σε κάθε επιτροπή και της έγκρισης των προτάσεων της Επιτροπής Γυναικών. Φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. Και όταν προσπαθούμε να διακριβώσουμε ποιος παράγον θα μπορούσε να επηρεάζει το ποσοστό έγκρισης των τροπολογιών και προτάσεων της Επιτροπής ΦΕΜ σε άλλες επιτροπές, προσπαθούμε να επαληθεύσουμε τρεις υποθέσεις. Η μία είναι ότι παίζει η ισορροπία των φίλων σε αυτή την Επιτροπή. Αν υπάρχει μεγαλύτερος αριθμό γυναικών, υπάρχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερο ποσοστό έγκρισης. Αλλά όπως είδαμε προηγουμένως, η σχέση αυτή δεν φαίνεται ιδιαίτερα εύρωστη. Από ό,τι φαίνεται από την ανάλυση μας, είναι πιο σημαντική η ικανότητα του κάθε εισηγητή από την παρουσία γυναικών για να υποστηριχθεί η έγκριση προτάσεων και τροπολογιών. Υπάρχει μια δεύτερη υπόθεση. Αν υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ της έγκρισης των προτάσεων αυτών που έχει να κάνει με πολιτικού χαρακτήρα συνάφεια μεταξύ της εισηγήτριας της Επιτροπής ΦΕΜ και του εισηγητή της εισηγήτριας στην άλλη Επιτροπή. Ούτε και αυτό δεν επαληθεύεται. Φαίνεται ότι όσο πιο πολλά, ότι όσο διαφορετικότερα ήταν τα κόμματα των εισηγητών, τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα έγκρισης. Η τελευταία ε, υπόθεση ήταν το πόσο σημαντικό ήταν το θέμα. Αν το θέμα είναι ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό στα μέσα ενημέρωσης και στην αντίληψη της κοινή γνώμης και αν συζητάτε ως θέμα φίλου, τότε πιο εύκολα περνάνε οι τροπολογίες αυτές για την ισότητα των φίλων να εγκριθούν. Επομένως, η σημαντικότητα του θέματος και το γεγονός ότι δεν αφορούν ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα, αυτό είναι πιο σημαντικό από η πολιτική συνάφεια ή οτιδήποτε άλλο. Και εδώ βλέπουμε πόσο ποσοστό από τις προτάσεις ενεκρίθησαν τελικά στις άλλες επιτροπές και πάλι βλέπετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό Έγκριση είναι για τα εργαλεία και την ε, ε, συμμετοχή. Ενώ τα θέματα της βίας των γυναικών δεν φαίνεται ότι οδηγούν σε τόσο μεγάλη έγκριση. Ούτε το σχολείο, ούτε η παιδεία, ούτε τα φροντιστήρια. Δεν εγκρίνονται λοιπόν αυτά τόσο πολύ. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί σας δείχνει πώς τα προεξάρχοντα θέματα είναι αυτά τα οποία έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με την έγκρισή τους. Βλέπουμε τώρα τις τροπολογίες στην περίοδο υποανάλυση. 177 τροπολογίες είχαν κατατεθεί για 27 εκθέσεις και προτάσεις. Οι περισσότερες αφορούσαν την Επιτροπή Απασχόλησης. Υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ της Επιτροπής Γυναικών και της Επιτροπής Απασχόλησης. Αν, βλέπουμε το, αν δούμε το ποσοστό έγκρισης, βλέπουμε ότι οι τροπολογίες για εισαγωγή της διάστασης του φύλου έχουν μεγαλύτερο ποσοστό έγκρισης από γενικά τις ε, προτάσεις και τις γνωμοδοτήσεις. Κυρίως από ό,τι φαίνεται γιατί δεν περιλαμβάνουν ριζοσπαστικές αλλαγές. Περιλαμβάνουν την είσοδο στα κείμενα της λέξεως γυναίκα. Και επομένως αυτό δεν είναι μια μεγάλη αλλαγή κατατίθενται κατευθείαν προς την οικία έκθεση και δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων. Είναι πιο αποτελεσματικές λοιπόν από τις γνωμοδοτήσεις γιατί είναι πιο σύντομες, υποβάλλονται πιο γρήγορα και αφορούν πάρα πολύ στενά καθορισμένα θέματα. Είναι λοιπόν μια σημαντική βελτίωση των εργαλείων που έχει η Επιτροπή Γυναικών για να υποστηρίξει την διάσταση του φίλου, Τα άλλα δύο πράγματα τα οποία έχουν γίνει στο διάστημα αυτό είναι οι εκθέσεις πρωτοβουλίας, οι ιδέες και οι διαδικασίες με δύο ή παραπάνω επιτροπές, όπως και στην περίπτωση των εκθέσεων πρωτοβουλίας, συνδέονται με θέματα τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με την ισότητα των φύλων και είναι σημαντικά για τη δημιουργήση μεγαλύτερης συνειδητοποίησης για θέματα τα οποία δεν βρίσκονται στην γενική αντίληψη όταν μιλάμε για την ισότητα των φύλων. Είναι σημαντικά λοιπόν για το mainstreaming γιατί υποδεικνύουν το μίσο που μπορεί να ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που εμπλέκει πολλές επιτροπές, πάνω από μια επιτροπή, η ΦΕΜ μαζί με την ΛΥΜΠΕ και την Τζούριν, είχαν ε, συνεργαστεί σε, στα πλαίσια της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας και αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό για να προωθηθεί η νομοθεσία και οι πράξεις από το Κοινοβούλιο που να περιέχουν μεγάλη εστίαση στο mainstream στην εισαγωγή της διάστασης του φύλου. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προωθηθούν στο δυνατόν περισσότερο. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι το έχω πέντε άλλων Agri, Budget, Libe και Envy. Και να δούμε τι κάνουν όταν δεν εμπλέκονται οι γυναίκες. Αν δίνουν κάποια προσοχή στην ισότητα του φίλου ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποια συνεισφορά από την Επιτροπή ΦΕΜ. Αυτό που βγήκε λοιπόν από την έρευνα είναι ότι όλες τους εκτός από την Επιτροπή Προϋπολογισμών αντιμετώπισαν τα θέματα αυτά κατευθείαν στο ίδιο τους το έργο. Αλλά, Αλλά... βλέποντας τα υπόλοιπα πράγματα που έκαναν, βλέπουμε ότι θα μπορούσαν να είχαν δώσει αυτή την προσοχή προς το, τη διάσταση του φίλου και σε άλλα θέματα που αντιμετώπισαν. Και εκεί λοιπόν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης η Επιτροπή ΑΦΕΤ είναι αυτή που δίνει μεγαλύτερη σημασία σε θέματα ισότητας των φύλων. Ένα 14%, των νομοθετημάτων τους αντιμετωπίζουν θέματα ισότητας των φύλων. Ακολουθεί η ΛΥΜΠΕ με 16% και η ΕΝΒΗ με 7,7%. Η Άγρη δεν έχει λάβει υπόψη τη θέση της γυναίκας αγρότησας και δεν έχει παραγάγει καμία ε, έκθεση που να έχει υπόψη τη την ισότητα του φίλων, αλλά πριν από λίγο καιρό είχαν μια σημαντική έκθεση για το ρόλο της αγρότησας στην αγροτική οικονομία. Δεν κάναν λοιπόν τίποτα περισσότερο. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών όμως μπορούσε με να αντιμετωπίσει θέματα ισότητας των φύλων, δεν το έπραξε δε. Είναι λοιπόν η Επιτροπή Προπολογισμών μια επιτροπή όπου είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να δοθεί περισσότερη σημασία στα θέματα αυτά. Και από την ανάλυση αυτών των πέντε επιτροπών εξάγεται ότι η σημαντικότητα του θέματος είναι πολύ σημαντικό συντελεστής. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουν κατευθείαν τα θέματα ισότητας των φύλων, είναι όταν τα θέματα αυτά βρίσκονται ήδη στα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες και ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη. Η ΑΦΕΤ παραδείγματος χάρη αντιμετωπίζει τα θέματα ανάπτυξης αντιμετωπίζει το θέμα της ισότητας των φύλων σε αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ένα πολύ γνωστό, πολύ συζητημένο ε, θέμα στην Ευρώπη. Και για να κλείσω, τι προτείνουμε, σε τι καταλήξαμε με αυτή τη μελέτη. Πρώτα απ' όλα είδαμε τη σημασία του ρόλου της Επιτροπής Γυναικών, τη σημασία της φήμης του της εισηγήτριας και το, τη σημασία τη σημαντικότητα του κάθε θέματο. Πώ θα βελτιώσουμε λοιπόν τα πράγματα αυτά για να κάνουμε τα θέματα αυτά ορατότερα, η Επιτροπή ΦΕΜ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της να προκαλεί συζήτηση και μέσα αλλά και έξω από το Κοινοβούλιο σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα ισότητας των φύλων, τα οποία συνήθω δεν αντιμετωπίζουν. Παραδείγματο χάρη, τα θέματα ισότητας των φύλων στον προπολογισμό. Μπορούμε να κάνουμε πολλά εκεί με το λεγόμενο gender budgeting, αλλά οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο προπολογισμό δεν έχει τίποτα να κάνει με την ισότητα των φύλων. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε δικέ μα εκθέσει πρωτοβουλία που θα αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε και να προωθήσουμε γεγονότα για το θέμα αυτό και να έχουμε επικοινωνία για τα θέματα αυτά μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα συμμετάσχουν στα θέματα αυτά ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τη σημασία της ισότητας των φύλων ακόμα και στα θέματα που τώρα δεν θεωρείται τόσο σημαντικό θέμα αυτό. Τώρα, για να αυξηθεί ο ρόλος των γυναικών στη λήψη αποφάσεων θα έπρεπε να δοθεί περισσότερη προσοχή στο θέμα του συντονισμού για να δούμε πότε μπορεί να συνδεθεί με άλλες επιτροπές για να πιέσει να προωθήσει τέτοια θέματα, να σχεδιάσει συνεργασία με άλλες επιτροπές για εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται κάποιος μηχανισμός πιθαναγκασμού, δηλαδή άμα σε βοηθήσω εγώ να με βοηθήσεις και εσύ, μεγαλύτερη συνεργασία και για να επιλεγούν καλύτερα τα θέματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γνωμοδοτήσεις, πολλές. Καλύτερο είναι να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε μερικές όπου να είμαστε πιο αποτελεσματικές. Και μετά οι τροπολογοί, οι συντάκτες τροπολογιών η σύνταξη τροπολογιών για θέματα ισότητας των φύλων να προωθείται και τέλος να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των οργάνων και δικτύων προώθησης ισότητας των φύλων χρειάζεται καλύτερο συντονισμός και αν είναι δυνατόν και εκπρόσωποι που προωθούν αυτά τα θέματα να συνεργάζονται περισσότερο με την Επιτροπή Γυναικών ή αν δεν είναι αυτό δυνατόν να ενδυναμώνονται οι σχέσεις μεταξύ των μελών της Επιτροπής Γυναικών και των εκπροσώπων της ισότητας των φύλων. Οι αξιολογήσεις τώρα θεωρούνται πολύ σημαντικό θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άρα μπορούμε να βάζουμε σε όλες τις αξιολογήσεις και το θέμα της ισότητας των γενών όταν νομοθετούμε να προωθούμε την ανάληψη μελετών με ιδιαίτερα με αυτό το εργαλείο Gender Impact Assessment που λέμε ώστε να βλέπουμε σε ποιες περιπτώσεις είναι σημαντικότερο να τίθεται το θέμα της ισότητας των φίλων. Η γραμματεία της Επιτροπής Γυναικών να μπορεί να βοηθάει τους ευρωβουλευτάς για να είναι πιο αποτελεσματική. Με συγχωρείτε γιατί μακρηγόρησα, αλλά να, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα μιλήσω σου ειδικά. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση που μας κάνατε. Okay, I continue with English and Dorian though, because I want to hear what is what I'm, I want you to hear what I'm saying. Φορέστε τα ακουστικά σας παρακαλώ για να καταλάβετε τι λέω. Νομίζω πως ε, ήταν πολύ σημαντικά τα όσα είπατε. Ε, πολύ ενδιαφέρον ε, ότι να βλέπουμε τέτοια ανάλυση της ίδιας της Επιτροπής. Μπορείς να τα μάθεις πάρα πολύ καλά για να δεις πώς κάποιος εκτός βλέπει τα πράγματα. Πολύτιμα τα στοιχεία που μας δίνετε. Να δούμε τι διδάγματα θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις, αλλά πρώτα θα έπρεπε να δώσω το λόγο στην κυρία Κορνέλισεν γιατί εκείνη ε, είχε την πρωτοβουλία για αυτή τη μελέτη και τώρα θα λέω σου ειδικά από εδώ και μπρος. Ε, jo, jag Το άκουσα και εγώ αυτό νωρίτερα, ότι κάποιες φορές κάνουμε εξαιρετικά πολλές γνωμοδοτήσεις. Το έχω ήδη ακούσει και καταλαβαίνω αυτό που εννοείται. Αλλά γιατί συντάσσουμε τόσε συνωμοδοτήσει, Αυτό είναι επειδή οι άλλε επιτροπέ ε, δεν τα πάνε καθόλου καλά όσον αφορά το mainstreaming και την, ε, το θέμα των γενών ή του φίλου. Και πρέπει λοιπόν κάθε φορά να παρέμβουμε για να διορθώσουμε τα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτό το μελετήσατε στη μελέτη σας. Εγώ πιστεύω πως τα σχόλιά μας λαμβάνονται υπόψη από τις επιτροπές που τα πάνε καλά όσον αφορά το mainstreaming. Είναι αυτές δηλαδή οι οποίες ε, δεν χρειάζεται να τις ε, να επιμείνουμε γιατί ήδη κάνουν την ε, δουλειά που πρέπει. Και επίσης είναι πιο ευαίσθητες όσον αφορά τη λήψη υπόψη, του, των τοπολογιών μας, διότι ήδη βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος Όμω με την Επιτροπή του προπολογισμού έχουμε μεγάλο πρόβλημα, διότι ας πούμε, το κείμενο της Ευρωπαϊκής Συνθήκη που λέει ότι όλες οι πολιτικές θα πρέπει να διέπονται από το mainstreaming του φύλου, εκεί χρειάζονται πόροι εφόσον θέλουμε πραγματικά να ανταποκριθούμε στο γράμμα των συνθήκων. Και έπειτα υπάρχει και το θέμα της ουδετερότητας των φύλων. Ε, μόνο που ο προπολογισμός δεν λειτουργεί έτσι. Και εκεί σίγουρα πρέπει να κάνουμε περισσότερα ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε τους εκπροσώπους του προπολογισμού να τους ευαισθητοποιήσουμε στα θέματα του φίλου. Η κυρία Κλειβέτη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικό που παραβρέθηκα σήμερα εδώ Ακόμα και αν έχει τυπωθεί βέβαια αυτή η μελέτη και βεβαίως θα τη μελετήσω προσεκτικά, ήταν πολύ σημαντικό να ακούσουμε άμεσα τα όσα είπατε εσείς. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελα να πω, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κυρίως άμεσα. Προσπαθείτε να κατανοήσετε ποιος είναι ο ρόλος των ανδρών στα θέματα του φίλου. Γιατί έχουμε άντρα πρόεδρο, που είναι καλό κατά τη γνώμη μου, αλλά κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο ρόλος ε, της συνεργασίας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση του θέματος της ισότητας των φύλων. Δεύτερον, είπατε ότι υπάρχουν ε, επιτροπές που ξεχνούν την διάσταση του φύλου και θεωρούν ότι τα θέματα αυτά είναι εκτός θέματος ενώ στην ε, πράξη θα έπρεπε να αναλύσουν τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν από την άποψη του φίλου αυτομάτως μάλιστα. Εσείς ε, μπορείτε να μας κάνετε κάποιες συστάσεις προς τις άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να μην ξεχνούν ότι υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα, σε όλες μάλλον τις αποφάσεις που λαμβάνουν και όλα τα θέματα που συζητούν. Υπάρχουν διαφορές και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Δεν ξέρω, ίσως να είναι κάπως υπερβολικά αυτά που λέω, αλλά σύντομα θα γίνουν οι εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο. Μπορείτε να λάβετε υπόψη ε, το θέμα αυτό και να στείλουμε ένα γράμμα στις πολιτικές, ε, στα πολιτικά κόμματα και τις πολιτικές ομάδες που να λένε σημειώστε και προσέξτε τη συμμετοχή των υποψηφίων που θα στείλετε. και να λάβετε υπόψη το θέμα του φίλου και εκεί, γιατί δυστυχώς πολύ λίγος κόσμος ενδιαφέρεται και ειδικεύεται για το θέμα του φίλου. πολλοί θεωρούν ότι «Ε, αυτά είναι τα θέματα των γυναικών και δεν δίνουν περισσότερη σημασία. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα τρει ε, στον κατάλογο των ομιλητών. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, γιατί έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα να εξετάσουμε. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Λούλινγκ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ζητώ συγγνώμη που έφτασα λίγο καθυστερημένα, αλλά είχα μια ομάδα επισκεπτών Άκουσα όμως ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της εισήγησης, της παρουσίασης και θα σας πω ότι εκπλήσωμαι. Γιατί είναι αστείο να φέρνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται άμεσα από το 79, να φέρνουμε κάποιον εδώ για να μας πει πώς πρέπει να οργανωθούμε. Εγώ είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής από τότε που πρωτοδημιουργήθηκε. Ήδη είχα υποβάλει ε, εκθέσεις, το 65 στην τότε Κοινωνική Επιτροπή είχα κάνει εκθέσεις, μια σύσταση μάλλον ήταν μόνο, για την προστασία της μητρότητας. Και θα πρέπει να σας πω ότι συμμετέχω και σε άλλες επιτροπές, όπως η Οικονομική και Νομισματική, η Επιτροπή της Γεωργίας. Είπατε ότι οι επιτροπές δεν λαμβάνουν υπόψη το φίλο. Μα δεν είναι αλήθεια αυτό. Εγώ θυμάμαι πολύ πρόσφατα Χάσαμε ώρες και ώρες στην Επιτροπή την Οικονομική και Νομισματική για να συζητήσουμε τη συμμετοχή ή τον ορισμό γυναικών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καθυστερήσαμε τον διορισμό του ε, διοικητή που ήταν μάλιστα και από τη χώρα μου επειδή δεν ήταν γυναίκα. Έχουμε κάνει λοιπόν φοβερά και δρομερά πράγματα. Είμαι και μέλος ε, της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Ε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει άριθμες εκθέσεις για την κατάσταση των αγροτισών. Και εγώ εδώ έχω κάνει πολλά αιτήματα και ψηφίσματα για την ισότητα μεταχείρισης ανδρών γυναικών και συζύγων ιδιαίτερα όσον αφορά τη γεωργία, ώστε να τη χάνουν τις ίδιες μεταχείρισεις. Μάλιστα πρόσφατα ε, συνέταξα μια έκθεση που έχει ήδη υιοθετηθεί για την ισότητα μεταχείρισης, όπου εδώ σε αυτήν εδώ την Επιτροπή καταφέραμε μαζί με το Σύμβουλο των Υπουργών να θεσπίσουμε τη δυνατότητα κοινωνικής ασφάλισης για τους συζύγους. Συζύγους. Ή τις, τους τις συζύγους, κυρίως στον τομέα της γεωργίας. Δηλαδή, δεν μας λέτε τίποτα το νέο. Δεν το ζήσατε εσείς αυτό βέβαια, αλλά πρέπει να σας πω ότι στην αρχή όταν φτιάχτηκε η Επιτροπή των Δικαιωμάτων της Γυναίκας, μπορέσαμε μια χαρά να ξέρουμε πού θα υποβάλουμε γνωμοδότηση. Ίσως να μην κάναμε τόσες πολλές εκθέσεις πρωτοβουλίες, γιατί τότε δεν ήταν της μόδας όπως είναι σήμερα. Αλλά το να λέει κανείς πως το Ευρωκοινοβούλιο, από τότε που υπάρχει, δεν έχει ασχοληθεί με τα δικαιώματα της γυναίκας, είναι ψέμα. Εγώ η ίδια έχω υποβάλει ένα σώρο εκθέσεις και, εκθέσεις και ψηφίσματα πρωτοβουλίας από το 65 για να προωθήσω την ισότητα μεταχείρισης, ισότητα μεταξύ των φύλων. Και δεν πρέπει να παρασταίνουμε ή να κάνουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασχολείται με την ισότητα των φύλων και από το, και από 75 γιατί εδώ θέλουμε να επενεφεύρουμε τον τροχό. Από το 75 Έχουμε 11 οδηγίες που αφορούν την ισότητα μεταχείρισης των γυναικών σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν κάποιες που χρειάζονται βελτίωση και μπορούμε να τη βελτιώσουμε αυτή που αφορά την προστασία της μητρότητας. Αν δεν είχαμε υιοθετήσει εδώ την έκθεση φουρτού που κανένα Συμβούλιο Υπουργών δεν θέλει να, το να τη συζητήσει, αν είχαμε εστιάσει στα όσα αφορούν την οδηγία περί προστασίας της μητρότητας θα είχαμε ήδη προχωρήσει πολύ περισσότερο. Έχουμε μια οδηγία για την ε, γονική άδεια. Έχουν συζητήσει για το θέμα αυτό οι κοινωνικοί εταίροι και επίσης και για την πατρική άδεια. Πρέπει να το προωθήσουμε. Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε λες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει συζητήσει τα θέματα αυτά. Αυτό είναι αστείο το 2014 να έχετε κάποιον που να μας λέει πώς θα πρέπει να οργανωθούμε. Ευχαριστώ, λέει κυρία Λούλιν. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι είπε κανένα ότι δεν υπήρχε πρόοδος. Η κυρία Χάνιμπολ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη γενική επισκόπηση που μας κάνατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη. Ελπίζω ότι θα μας διανεμηθεί και σε έγγραφη μορφή, γιατί είναι ένα πολύ χρήσιμο έγγραφο για μας. Συζητάμε στην Επιτροπή αυτή για την εισαγωγή της διάστασης του φίλου για πάρα πολύ καιρό. Έχει δίκιο η κυρία Λούλιν. Αυτό που έδειξε η έκθεσή σας είναι ότι έχουμε κάνει πρόοδο. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Αλλά δεν έχουμε πετύχει αυτό το οποίο θέλουμε. Δεν έχουμε πραγματικά αντιμετωπίσει τη συνολική αυτή πρόκληση. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία φυσικά συνδέονται με την ε, απασχόληση, αλλά ήταν ενδιαφέρον αυτό που βρήκατε ότι πράγματι εκεί είναι η μεγαλύτερη αιστείας δεδομένου του τι κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι λιγάκι αναπόφευκτο να υπάρχει τόσο μεγάλη έμφαση στην ισότητα σε θέματα απασχόλησης. Αυτό το οποίο με στενοχώρησε τώρα και με σεκλέτησε είναι το εξής. Ότι το μήνυμά μας δεν περνάει. Ίσως θα πρέπει να ξεπεράσουμε το στενοκύκλο της Επιτροπής. Και όπως είπε και η ομιλήτριά μας, έχουμε προχωρήσει, αλλά δεν έχουμε μπει στον πυρήνα των πραγμάτων. Και δεν έχουμε κάνει όλα αυτά πρέπει να κάνουμε. Αναρωτιέμαι, πού μπαίνει τώρα, πού κολλάει η συνέλευση των Προέδρων. Μήπως θα πρέπει να φέρουμε ορισμένα θέματα στη συνέλευση των Προέδρων για να τα αντιμετωπίσουν και αυτοί στο δικό τους επίπεδο. Και επίσης θα συζητηθεί και σε επίπεδο πολιτικών ομάδων. Γιατί υπάρχουν κάποια επίπεδα της οργάνωσης τα οποία δεν αναφέρονται στην έκθεση και προφανώς κάτι γίνεται εκεί. Αλλά πιστεύω για την επόμενη θητεία Ίσως θα μπορέσαμε να βρούμε μια στρατηγική για να συνεχίσουμε την πρόθεση των θεμάτων ισότητος. Όλα αυτά που κάναμε ήταν καλά, αλλά ήταν λιγάκι ασύνδετα. Σίγουρα πρέπει να δούμε τι γίνεται στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Και θα ήταν χρήσιμο να μην αφήσουμε αυτή την έκθεση απλώς να μπει στο αρχείο, αλλά να προχωρήσουμε επί τη βάση των πολύ καλών προτάσεών της για να καταλήξουμε και εμείς σε κάποιες κοινέ θέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να προσθέσω και εγώ τις ευχαριστίες μου σε αυτές των συναδέλφων που εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το τόσο σημαντικό αυτό έργο ερευνητικό και το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και εύστοχο διότι η οπτική γωνία των ε, εμπειρογνωμόνων είναι συμπληρωματική με αυτή των πολιτικών και μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα την πραγματικότητα. Ο καθένας έχει το δικό του λόγο, λόγο και ρόλο σε αυτόν τον πολύπλοκο κόσμο που λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις. Πιστεύω ότι έγινε σαφές και από αυτή τη μελέτη ότι ακόμα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα νοοτροπίας. Υπάρχουν τα στερεότυπα ή προκαταλήψεις, ακόμα και σε επίπεδο πολιτικού λόγου. Η συμπερίληψη της ισότητας των φύλων χρησιμοποιείται μόνο περισσότερο για εκλογική εκμετάλλευση. Γιατί αυτό φυσικά είναι ένα σύνθημα που είναι πολιτικά ορθό και οι πολιτικοί το κάνουν για αυτό το λόγο, αλλά δεν το κάνουν επειδή είναι πεπισμένοι για την ανάγκη ισότητας των φύλων. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε στην πράξη, όπου δεν υπάρχει πραγματικά σχέση αιτίου και αποτελέσματος μεταξύ των λόγων και αυτών που γίνονται στην πράξη. Σε σχέση με τη μελέτη αυτή καθεαυτή και τα ερωτήματα που θα είχα εγώ να κάνω σε σχέση με τη μελέτη αυτή, νομίζω ότι αλλά με υπόψη το πλαίσιο κρίσης στο οποίο βρισκόμαστε, το οποίο έχει οξύνει τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και σε επίπεδο λοιπόν απασχόλησης και σε επίπεδο ψαλίδας αποδοχών που έχει ανοίξει ακόμα περισσότερο, θα ήθελα να θέσω το ερώτημα του κατά πόσο από τη δική σας εμπειρία στις μελέτες που έχετε κάνει στο παρελθόν και σε αυτή τη μελέτη προκύπτει ότι υπάρχουν αρνητικές συνέπειες από την κρίση σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων. Και η άλλη ερώτηση που ήθελα να θέσω είναι η Μέχρι ποιου σημείου μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι υπάρχει μικρότερη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, ακόμα και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών οργάνων, ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αν αυτό έχει κάποιες συνέπειες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίμα που έφυγε η κυρία Λούλινγκ. Γιατί ήρθε χωρίς να έχει ακούσει την παρουσίαση της μελέτης, ούτε έμεινε να ακούσει τα σχόλια των άλλων βουλευτών. Δεν μας ακούει. Και είναι κρίμα λοιπόν πρέπει να αναφερθώ και στο σημείο αυτό ότι δεν βοηθάει καθόλου σε σχέση με την προβληματική των δικαιωμάτων των γυναικών να υπάρχουν γυναίκες οι οποίες χρησιμοποιούν τη μεγάλη τους πείρα και ικανότητα για να στρέφονται κατά άλλων γυναικών και κατά της Επιτροπής μας η οποία ανέκρινε σημαντικές εκθέσεις, στη δική μου έκθεση για την αναθεώρηση της οδηγίας για την μητρική άδεια που ενεκρίθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία και πιστεύω ότι είναι μια σαφής πρόταση και ακόμα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προ του οποίου κύπτουν τον αυχένα πάρα πολύ ακόμα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο έχει άλλες προτεραιότητες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτό είχε μια θέση η οποία ήταν μερκαντιλιστικού χαρακτήρα, εμπορικού χαρακτήρα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζούμε. Πρέπει λοιπόν σαν αντίβαρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μια πιο κοινωνική αντιμετώπιση για τα δύο φύλλα, για τις γυναίκες και τα παιδιά. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι ως γυναίκα και ως αντιπρόεδρος αυτής της Επιτροπής πρέπει να εκφράσω την ε, δυσαρέσκειά μου γιατί υπάρχουν γυναίκες οι οποίες μας κατηγορούν περισσότερο από ότι οι άνδρες. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Μπορούμε να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στην ομιλήτριά μας για να δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Σύντομα όμως γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ. Yes, just few words. Ε, first... Ε, ναι, δύο λόγια μόνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το gender mainstreaming και το όσα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των ετών στο Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο προηγμένα θεσμικά όργανα στα θέματα αυτά. Αυτό που κάναμε δεν ήταν να πούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει, ε, υπάρχει μάλιστα ένα ολόκληρο κεφάλαιο που λέει το τι έχει γίνει και αναγνωρίζει τη σημασία του Κοινοβουλίου για το gender mainstreaming. Αυτό που κάναμε ήταν να δώσουμε ε, έξωθεν να δείξουμε κάποια κρίσιμα ζητήματα που θα μπορούσαν να εξεταστούν ώστε να αυξηθεί, να βελτιωθεί, να βελτιωθεί η κατάσταση ακόμη περισσότερο. Θελήσαμε λοιπόν να εξετάσουμε ορισμένα θέματα εμείς, τα υπόλοιπα εσείς θα τα αποφασίσετε τι πρέπει να κάνετε. Αν αυτά που σας δώσαμε σας σωθούν να είστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτά που είπα στο τέλος λοιπόν είναι απλώς ένας κατάλογος θεμάτων και μερικές συστάσεις και θα τις συζητήσετε και θα δείτε πώς να συνεχίσετε. Ένα από τα θέματα ήταν ότι θέλαμε να είμαστε πιο επιλεκτικοί γιατί θέματα ισότητας των φύλων σε μερικούς τομείς είναι γνωστά, σε άλλους όχι. Λόγω λοιπόν των πολιτήμων ανθρωπίνων πόρων που διαθέτεται, παρά το ότι τους διαθέτεται δεν μπορείτε να τα κάνετε και να τα παρακολουθήσετε όλα. Χρειάζεται λοιπόν κάποια επιλογή και θα ήταν σωστό να συνεχίσουμε έτσι με μια, τον καθορισμό κάποια στρατηγικής. Η επικοινωνία επίσης είναι πολύ σημαντική για να δείξουμε προς τα έξω τι κάνουμε. Είδαμε ποια είναι η δραστηριότητα των μέσων μέσα στο Κοινοβούλιο για τα θέματα ισότητας των φύλων και δεν είναι και τόσο μεγάλη. Δεν είναι πολύ ορατό το θέμα στα μέσα. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσατε να προωθήσετε. Τώρα ο ρόλος των ανδρών και αυτός είναι σημαντικός, ε, σημαντικός. Γιατί είναι όλο και σαφέστερο ότι αν θέλουμε να αυξήσουμε την ανάπτυξη στην Ευρώπη χρειάζονται περισσότερες γυναίκες να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Γιατί το μισό πληθυσμό δεν τον απασχολούμε για αυτόν τον στόχο και είναι ο μισός πληθυσμός που τώρα έχει πολύ καλή εκπαίδευση και παιδεία και άρα πρόκειται για κατασπατάληση ανθρωπίνων πόρων. Η κρίση τώρα. Μέχρι τώρα επλήγησαν περισσότερο οι άντρες παρά οι γυναίκες από την κρίση. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος όλες οι υπηρεσίες τελικά να αναλυφθούν από να αναλάβουν το βάρος οι γυναίκες της κρίσης γιατί θα γίνουν μειώσεις θέσεων, απολύσεις. Η πολιτική εκπροσώπηση επίσης. Στην Ιταλία πριν από μερικές μέρες το η Βουλή καταψήφισε ένα εργαλείο προώθησης της ισότητας των φύλων στην προετοιμασία των εκλογικών καταλόγων και επομένως όλα τα κόμματα, οι άντρες από όλα τα κόμματα το καταψήφισαν. Αυτά είναι σημαντικά και για τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να υπάρχει ένα εργαλείο που να εγγυάται την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ρόλος της διάσκεψης των προέδρων κλπ. Υπάρχουν μερικές συστάσεις στην έκθεση και που τις θεωρούμε σημαντικές. Το ότι εσείς έχετε άντρα ως πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών είναι καλό, διότι είναι πιο αποδεκτός από τους άλλους. Δυστυχώς ακόμα εκεί βρισκόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι τα καταφέρατε πολύ καλά και ελπίζω και στην επόμενη θητεία να συνεχίσετε σε αυτόν τον δρόμο και να μπορέσετε να συνεχίσετε το έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Σας κατευχαριστούμε για τις πολυτιμότατες αυτές πληροφορίες και συμβουλές. Έχω διαβάσει τη μελέτη και ε, την εκτιμώ ιδιαίτερα. Δυστυχώς βέβαια οι άντρες ακούνε περισσότερο άλλους άντρες και όχι τις γυναίκες. Αυτό είναι κρίμα. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι τη μελέτη τη ζήτησε το τμήμα κατάστρωσης πολιτικής και αφορούσε κυρίως την αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας της Επιτροπής ΓΙΝ. Η κυρία Κορνέλησεν την είχε πρωτοζητήσει. Και γι' αυτό καταλήξαμε τελικά να σας έχουμε εδώ. Είναι πολύ καλό κάποιος εκτός του Κοινοβουλίου να κάνει αυτές τις μελέτες. Φυσικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούσαμε και η μελέτη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Συνεχίζουμε τώρα στο 1. τα δημογραφικά θέματα που έθεσε ο ΙΕ θα μας κάνει μια παρουσίαση η αρμόδια διευθύντρια του ΟΗΕ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία σας. Έχετε βέβαια μόνο 10 λεπτά, αλλά είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που σας βλέπουμε, γιατί και η δική σας δουλειά σχετίζεται με τη δική μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Την άδελφη. 600 εκατομμύρια γυναικών και κοριτσιών ζουν σε, σε χώρε. χώρες. Οι δυνατότητες που έχουν κατά την εφηβεία τους θα καθορίσουν κατά πόσο θα αρχίσουν να δουλεύουν ως ε, ισότιμοι πολίτες με όλες τις δυνατότητες που μπορούν να έχουν. Αλλά οι πρώιμες εγκυμοσύνες συχνά υπονομεύουν τις δυνατότητες αυτές και δεν έχουν έτσι το μέλλον που θα μπορούσαν να έχουν. Γι' αυτό ο οργανισμός μας έκανε μία μελέτη, μία αναφορά το 2013 με τίτλο «Μητρότητα και παιδική ηλικία» και τονίζει τους κινδύνους της εφηβικής εγκυμοσύνης. Επίσης έδειχνε τι μπορούσε να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Τον περασμένο μήνα επίσης κάναμε την έκθεση ICPD πέρα από το 2014 που ε, αξιολογούσε την πρόοδο, τα, τις ελλείψεις, τις προκλήσεις σχετικά με το πρόγραμμα δράσης που είχε εγκριθεί στο Κάιρο πριν από 20 χρόνια. Στη σημερινή μου παρουσίαση θα συγκεντρωθώ στα θέματα της εφηβικής εγκυμοσύνης με βάση τις συστάσεις και τα συμπεράσματα και από τις δύο αυτές εκθέσεις. Η μητρότητα στην παιδική ηλικία είναι πρόβλημα. Ποια είναι τα στοιχεία. Στι αναπτυσσόμενε χώρε κάθε χρόνο 7,3 εκατομμύρια κορίτσια κάτω των 18 ετών γεννούν. Από αυτά τα 7,3 εκατομμύρια κορίτσια, 2 εκατομμύρια είναι κάτω των 15 ετών και 90% των γενών γίνονται με γάμο. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά σχετίζονται με τους παιδικούς γάμους που βία φέρνουν στην ε, ενήλικη περίοδο τα νεαρά κορίτσια. Παρά το ότι είναι ακόμη παιδιά. Αν συνεχίσει η ίδια τάση μέχρι το 2020 142 εκατομμύρια κορίτσια θα, παντρεύουν, θα είναι ήδη παντρεμένα μέχρι το 18 τους. Σε όλες τις περιοχές του κόσμου οι αγρότησες ε, είναι εκείνες που κυρίως εγκυμονούν νωρίτερα. Επίσης κορίτσια από εθνοτικές μειονότητες ή περιθωριακές ομάδες και που δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση για την αναπαραγωγή. Και η έκθεση αυτή καταλήγει ότι η εφηβική εγκυμοσύνη είναι πολύ μεγαλύτερη πρόκληση στον αναπτυσσόμενο κόσμο παρά στον αναπτυγμένο. Και ότι επίσης στις αναπτυγμένες χώρες 680.000 γεννήσεις ε, εφήβων συμβαίνουν παρόλα αυτά κάθε χρόνο. Στον χάρτη αυτόν βλέπετε το ποσοστό γυναικών 20 με 24 που έχουν γεννήσει πριν τα 18. Επίσης βλέπετε ότι το ποσοστό είναι μεγαλύτερο στις χώρες που είναι με κόκκινο και λίγο χαμηλότερο πορτοκαλί. Δηλαδή στην υποσαχάρια Αφρική και την Νότια Ασία. Το κίτρινο δείχνει ότι 10 με 20% των κοριτσιών κάτω από 18 εγκυμονούν και το μπλε κάτω από 10. Και το γκρι σημαίνει δεν έχουμε στοιχεία. Για να δούμε τώρα ποια αποτελέσματα έχει η φυσική εγκυμοσύνη. Όταν ένα κορίτσι εγκυμονεί ή γεννάει, η υποβαθμίζονται όλες τις δυνατότητες για μελλοντική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Οι επιπτώσεις στη νεαρή μητέρα συνήθως ε, μεταφέρονται και στο παιδί της που αρχίζει τη ζωή με υποβαθμισμένες δυνατότητες. Το κόστος επίσης της εφηβικής εγκυμοσύνης ξεπερνάει μόνο τα συμφέροντα της ίδιας της νεαρής μητέρας, αλλά αφορά όλη της την οικογένεια και κοινότητα και την οικονομία της χώρας της. Υπάρχει επίσης πολύ μεγάλη υγειονομική επίπτωση και για τη μητέρα και για το παιδί. Γιατί πολλές φορές τα κορίτσια 15 με 19 που γεννούν ε, καταλήγουν στο θάνατο. 70.000 έφηβες πεθαίνουν κάθε χρόνο για λόγους που σχετίζονται με εγκυμοσύνη. Αυτό είναι τραγικό γιατί πολλά από αυτά, όλα από αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Επίσης πολλά ατυχήματα συμβαίνουν κατά τη γέννα, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική και την Νότια Ασία. Κορίτσια 15 με 19 ετών υφίστανται 3,2 εκατομμύρια εκτρώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης πολλές φορές ε, έχουν πολύ κακή διατροφή Μία, στις, μία, ένα στα δύο αυτά κορίτσια έχουν ανεμία και αυτό μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο της πρόορης γένας. Η ε, θάνατη των νεογέννητων είναι κατά 50% υψηλότερη μεταξύ των παιδιών από έφηβες μητέρες. Όταν φτάνουν την εφηβεία τα κορίτσια, οι ανάγκες τους για σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία αυξάνονται. Το να υπάρχει πρόσβαση σε αμερόληπτη πληροφορία είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα κορίτσια. Η πρόορη η εγκυμοσύνη έχει και επίπτωση στην εκπαίδευσή τους. Για πολλές κοπέλες φύγεται η δυνατότητα παιδείας τους αναγκάζονται να φύγουν από το σχολείο λόγω πιέσεων της κοινότητας ή λόγω του γεγονότος ότι τα σχολεία δεν επιτρέπουν στα έγκυα κορίτσια να πηγαίνουν σχολείο ή να ξαναγυρίσουν όταν γυρίσουν. Ακόμα και σε χώρες όπου υπάρχει δυνατότητα να γυρίσουν, πολύ λίγες κοπέλες επανέρχονται στην παιδεία. Όσο περισσότερο μένει εκτός σχολείου ένα κορίτσι και τα αγόρια το ίδιο, το λιγότερο πιθανό που είναι να ξαναγυρίσουν. Από την άλλη πλευρά, τα κόρυφα που μένουν περισσότερο στο σχολείο είναι πιο απίθανο να μην είναι έγκυες, γιατί η παιδεία προετοιμάζει τις γυναίκες για τις δουλειές της, αυξάνει την ε, αυτοεκτίμησή τους και το στάτους τους και τους δίνει περισσότερη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τις γονείς τους. Η παιδεία μειώνει τη δυνατότητα, την πιθανότητα να παντρευτεί ένα κορίτσι μικρό και καθυστερεί την γένα. Η χαμηλότερη ε, χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης συμβάλλει σε ε, υψηλότερη μάλλον εκπαίδευση βοηθάει να είναι και πιο υγιή τα μωρά. Υπάρχει και μια διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πρόορια εγκυμοσύνη. Γενικά υπάρχει πρόοδος προς την ισότητα των φύλων, αλλά σε πολλές περιοχές του κόσμου περιορίζονται επίτηδες τα δικαιώματα των γυναικών. Πουθενά δεν έχουν την ίδια οικονομική δύναμη με τους άλλους. Παρά την νομοθεσία εναντίον των αρνητικών πρακτικών, η γάμι παιδιών και ο ακροτηριασμός των γυναικείων ε, γεννητικών οργάνων παραμένουν σε πάρα πολλές χώρες. Το 2010, 158 χώρες είχαν ηλικία γάμου 18 ετών, αλλά το 1 τρίτο γυναικών που είναι τώρα 20 με 24 στις αναπτυσσόμενες χώρες, είπαν ότι είχαν παντευτεί, ήταν σε μια σταθερή σχέση πριν από τα 18 και 12 ήδη πριν από τα 15 τους. Μία στις τρεις γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο αναφέρει ότι έχει αντιμετωπίσει σωματική σεξουαλική βία, κυρίως στα χέρια ενός γνωστού και οικείου ατόμου. Η βία επί του φύλου είναι μια από τις πιο συνηθισμένε μορφές παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό οδηγεί σε μια ε, ανασφάλεια σε όλη τη διάρκεια τη ζωή για τι κοπέλε και τι γυναίκε. Αν μια κοπέλα δεν μπορεί να πάει στο σχολείο για την ή πρέπει να φροντίσει τα παιδιά τη χάνει τα δικαιώματά τη. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η αυτονομία της και η δυνατότητά της να έχει εισόδημα στη ζωή της και παραμένει εγκλωβισμένη στην ένδυα. Το να αντιμετωπίσουν λοιπόν την, ε, τις εγκυμοσύνες των εφήβων με ε, <clears throat> τρόπο που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα απαιτεί ένα διεθνές καθοριστικό, κανονιστικό πλαίσιο που θα σημαίνει ότι οι κυβερνήσει θα πρέπει να δώσουν στι κοπέλε τη δυνατότητα να ζήσουν ελεύθερε από βία και να έχουν τα δικαιώματα για υγεία και παιδεία. Τέλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει και οικονομική, οικονομικό αντίκτυπο τη της εγκυμοσύνης μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα για την παιδεία τους και την απόκτηση εισοδήματο. Αλλά το οικονομικό, δεν είναι μοναχα οικονομικό κόστος για αλλά και για όλη την κοινωνία και τη χώρα που βρίσκονται. Καταρχήν είναι μεγαλύτερη πίεση στα συστήματα α, περίθαλψης λόγω των ε, αμβλώσεων που πολλές φορές προκύπτουν. Αντίθετα, οι επενδύσεις οι οποίες δίνουν στις κοπέλες δυνατότητες να συμμετέχουν φέρνουν μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα για όλους. Η καθυστέρηση της γένας ε, δίνουν περισσότερες δυνατότητες στις γυναίκες για να αποκτήσουν κάποιο εισόδημα και βοηθούν την υγεία τους, την υγεία των οικογενειών τους και την γενικότερη υγεία γενικά. Οι επενδύσεις λοιπόν αυτές βοηθούν τη γενικότερη οικονομία και το κόστος της μη επένδυσης είναι πάρα πολύ μεγάλο άμα σκεφτεί κανείς το ευκαιριακό κόστος που έχει να κάνει με την ε, εγκυμοσύνη και το γεγονός ότι χάνουν το εισόδημα που θα μπορούσαν να αποκτήσουν αλλιώς οι γυναίκες αυτές. Τι πρέπει να γίνει τώρα με τις έφηβες κοπέλες. Μία ολιστική προσέγγιση απαιτείται για να, βελτιώσουν, να βελτιώσουμε τη ζωή αυτών των κορίτσιων. Πρέπει να υπάρχουν νόμοι οι οποίοι φέρνουν την ηλικία γάμου στα 18 και να προωθούν ε, προσπάθειες που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών και εμποδίζουν τους γάμους παιδιών. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση στην παιδεία των κοριτσιών. Θα πρέπει να έχουν σεξουαλική εκπαίδευση οι νέες κοπέλες για να αποκτήσουν τις ε, δεξιότητες που χρειάζονται για να προστατεύσουν την υγεία τους. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Χρειαζόμαστε καλής ποιότητας αναπαραγωγική υγεία που να είναι κατάλληλη για τα έφηβα κορίτσια και αγόρια ώστε να πάρουν τις σωστές επιλογές. Αυτό σημαίνει να εκπαιδεύσουμε τους παρόχους υγειονομικών υπηρεσιών ώστε να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των έφηβων κοριτσιών, ώστε να φύγει το στίγμα και ο φόβος που μαστίζει τις κοπέλες αυτές. Χρειαζόμαστε επίση μέτρα για να γίνουν πιο αυτόνομε αυτέ οι κοπέλε, για να αλλάξει η νοοτροπία για του ρόλου των φίλων και την ισότητα των φίλων και να εμποδίσουμε τη σεξουαλική βία. Κάτω από όλα αυτά βρίσκεται και η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προστασία της αξιοπρέπειας των νέων κοριτσιών. Πολλές φορές η κοινωνία είτε έμεσα είτε άμεσα λέει ότι το κορίτσι φταίει που έπνε έγκυος. Ενώ αυτό δεν γίνεται σε σαν αποτέλεσμα μιας απειλεγής, αλλά λόγω της έλλειψης επιλογών και συνθήκων που είναι πέρα από τον έλεγχο του κοριτσιού αυτού. Όπως σας είπα προηγουμένως, η εκθεσιά ICP την 2014 έκθεση επισκοπεί και αναδυθεί την πρόοδο, τα χάσματα και τις προκλήσεις σε σχέση με τις ε, περιπτώσεις αυτές που συνελέγει στη Διεθνή Συνδιάσκεψη του 1994 με στοιχεία από 176 χώρες και συμπηλεί τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και τις συνεισφορές της κοινωνίας των πολιτών και των ακαδημαϊκών. Ε, έχουμε την έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την παγκόσμια αυτή έκθεση ICPD. Την μπορείτε να τη βρείτε στην είσοδο στο τραπέζι. Η έκθεση αυτή θα συζητηθεί και στην Επιτροπή για το Πληθυσμό και την Ανάπτυξη που θα γίνει τον Απρίλιο. Τώρα, επειδή δεν έχουμε αρκετό χρόνο, δεν θα μπω σε όλες τις διάφορες συστάσεις και πορίσματα. Ένα σημαντικό θέμα είναι όμως ότι τα πορίσματα της έκθεσης σηματοδοτούν ε, τεράστια πρόοδο σε ορισμένους τομείς. Ένας εξ αυτών είναι η μείωση της στόχης που σημαίνει ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε απόλυτη φτώχεια έχει μειωθεί στο μισό, αλλά σε άλλες περιοχές τα προβλήματα και οι υποσχέσεις δεν υλοποιήθηκαν και ακόμα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Και αυτά νομίζω θα χαρείτε, γιατί τελείωσα την ε, εισήγησή μου με αυτή την παρατήρηση το πρόγραμμα δράσης, και αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της έκθεσης, συνέβαλε το πρόγραμμα ICPD σε απτή πρόοδο για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Λιγότερες γυναίκες πεθαίνουν ε, κατά την, τον τοκετό, περισσότερα κορίτσια έχουν πρόσβαση στην παιδεία και, στη, και πηγαίνουν στο σχολείο. Όμω, οι επιτυχίες δεν είναι ίσες για όλους. Στις στοχότερες κοινότητε, ακόμα και σε πιο πλούσιες χώρες, η θάνατος της μητέρας, η εφηβική εγκυμοσύνη και γενικά η πρόοδο ε, των ε, γυναικών ε, δεν είναι πολύ μεγάλη από το 1994. Αυτό που προκύπτει είναι ότι τα κέρδη αυτά δεν μπορούν να σταθεροποιηθούν ή να αυξηθούν αν δεν αντιμετωπιστεί η ανισότητα και οι διακρίσεις που είναι το χειρότερο. Είναι κρίσιμη η χρονιά αυτή εδώ για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη, για την χειραφέτηση των γυναικών και αυτά όλα στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας αναπτυξιακής ατζέντα, η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι οι κυβερνήσεις, κοινοβούλια, Ευρωπαϊκή Ένωση, ο και ΜΚΟ, είναι το πώς θα συνεργαστούμε μαζί ώστε να προστατευθούν και να προωθηθούν η ατζέντα της ε, χειραφέτησης των γυναικών ώστε να ενταχθεί στο πλαίσιο για μετά το 2015. Οι κυβερνήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο για την αναθεώρηση της ατζέντα στο ICPD και θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να ε, ενταχθούν όλα αυτά στην αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015 και την Ειδική Σύνοδο του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Εάν συνεργαστούμε μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα σεξουαλικά και τα παραγωγικά δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των εφήβων και των νέων, η ε, πάλιψη των διακρίσεων να θεωρηθούν ως σημεία κλειδιά για την ατζέντα μετά το 2015. Και κλείνοντας, ε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι μετά και πόσον είναι η τελευταία συνεδρία σε αυτή τη θητεία για την Επιτροπή σα, ότι εν μέρει χάρη στη σκληρή δουλειά του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας ε, η χειραφέτηση των γυναικών παραμένει ψηλά στην ημερήσια διάταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, βεβαίως και εμείς έχουμε ασχοληθεί με τις διεθνείς ε, σχέσεις. Είμαστε ευτυχείς που είστε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισήγησή σας. Ε, ε, ε, κυρία Μορβάη έχει ζητήσει τον λόγο. Θα σας δώσω μάξιμουμ δύο λεπτά, γιατί έχουμε και άλλη μια ομιλήτρια. Μάξιμουμ δύο λεπτά, παρακαλώ. Είναι λίγοι οι βουλευτές οι οποίες είναι παρόντες και δεν με εντυπωσιάζει το ότι έχουμε πίεση χρόνου, αλλά όταν έχουμε μία εκπρόσωπο του ΟΗΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία μας αναφέρει τα προβλήματα της, ε, της ε, πρόορης ε, εγκυμοσύνης, τι ε, κακή εντύπωση κάνουμε. Εμείς ασχολούμαστε μονάχα με τον τρίτο κόσμο αλλά δεν λέμε ότι το φαινόμενο αυτό έχει γίνει μαζικό και στην Δυτική Ευρώπη. Και επίσης ακόμα πιο έντονο έχει γίνει σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως στην Ουγγαρία, όπου μεταξύ του πληθυσμού των Ρωμά αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο. Όλα αυτά όμως είναι μια μορφή διάκρισης. Εσείς θέλετε να υποστηρίξετε την υγεία μια κοπέλα στην Αφρική και όχι μια κοπέλα Ρωμά στην Ουγγαρία. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Υπάρχουν σχετικά λοιπόν κάποιε έρευνε πώ μπορούμε να να εξασφαλίσουμε οι κοπέλες στο Ρωμά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά και να μάθουν να εκπαιδεύονται και να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να εξασφαλίσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους και να τη μεταλαμβαδεύσουν στην επόμενη γενιά και όχι να έχει μια γυναίκα 18 παιδιά και η επόμενη γενιά να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να συνεχίσω στο σημείο αυτό. Προφανώς αυτό δεν έχει να κάνει μονάχα με τον αναπτυσσόμενο χώρο. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα με εφηβικές εγκυμοσύνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να πω κάτι για το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι ίσως από τα χειρότερα παραδείγματα. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και βελτιώθηκαν και το έγινε αυτό γιατί υπήρξε μια παρέμβαση της κυβέρνησης. Το 1998 φτιάξαμε μια μονάδα κατά της, του κοινωνικού αποκλεισμού και το ένα πράγμα που αντιμετώπισε είναι οι ε, εφηβικές εγκυμοσύνες και η αντισύλληψη για τις νέες κοπέλες και έτσι μπόρεσε να μειώσει σημαντικά κατά πάνω από 40% τον αριθμό των εφηβικών εγκυμοσύνων που δείχνει ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης μπορεί πράγματι να λειτουργήσει αν υπάρξει πραγματική δραστηριότητα και αυτό έγινε από κοινού με τις τοπικές αρχές και τις υγειονομικές υπηρεσίες και φυσικά με εκπαιδευτικά ιδρύματα για να εξασφαλίσουμε ότι οι νέες αυτές κοπέλες παρέμειναν στο σχολείο και μετά βγαίναν στο χώρο εργασίας. Όλο αυτό το πρόγραμμα ήταν πολύ επιτυχημένο και είχε σημαντικό αντίκτυπο. Απλώς θέλω να το τονίσω αυτό ότι είναι ένα παράδειγμα του τι μπορεί να γίνει. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό ακόμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αλλά έχουν μειωθεί. Τα ποσοστά αυτά δεν είναι λοιπόν μονάχα ένα πρόβλημα του αναπτυσσόμενου χώρου, κόσμου, αλλά υπάρχουν λύσεις. Θα δώσω στην ομιλήτρια τώρα τη δυνατότητα να απαντήσει. Και ένα από τα σημαντικά πράγματα είναι ο νέος αυτός φορέας ο οποίος θα πρέπει να προωθήσει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πρέπει να υπάρξει μια οικουμενική αντιμετώπιση στα θέματα αυτά. Δεν είναι πρόβλημα λοιπόν στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι παντού σε όλο τον κόσμο. Έχετε το λόγο μου, τώρα. Πάρα πολύ σύντομα, σας ευχαριστώ. Για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι μίλησα πολύ γρήγορα. Μου το έπανε και οι διερμηνείς. Αλλά αυτό που ήθελα να πω να υπογραμμίσω είναι ότι όντω δεν είναι μόνο στι αναπτυσσόμενε χώρε πρόβλημα η εφηβική εγκυμοσύνη. Είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα εκεί, αλλά και στι βιομηχανοποιημένε χώρε υπάρχουν 600.000 και βάλε κορίτσια που γεννούν κάθε χρόνο. Ε, ε, σωστά το είπατε κι εσείς. Και το άλλο που ήθελα να πω και που αναφέρεται στην παγκόσμια έκθεση ε, ότι αυτό έχει να κάνει με την ανισότητα Ορισμένες ομάδες μπορεί να περιθωριοποιηθούν σε μια κοινωνία και βρίσκονται σε πολύ χειρότερη κατάσταση όσον αφορά τα σεξουαλικά αναπαραγωγικά δικαιώματα ή την εφηβική εγκυμοσύνη, αλλά μπορεί αυτό να μένει κρυφό γιατί ακριβώς ε, δεν τους λαμβάνει κανείς υπόψη. Φυσικά για τον ΟΗΕ, για το Ταμείο του Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών ε, ε, ασχολούμαστε με το θέμα, τα ξέρουμε ότι γίνεται αυτό και ότι υπάρχει αυτό. Και φυσικά η κατάσταση αυτή δεν είναι μοίρα, δεν είναι, μη δεν είναι το πεπρωμένο. Και οι δημόσιες πολιτικές όντως κάνουν τη διαφορά. Και οι δημόσιες πολιτικές που δεν έχουν στόχο μόνο τις γυναίκες, τα κορίτσια που τους λένε ναι, ότι δεν είναι καλό να μένετε έγκυες τόσο νέες, αλλά που αναντιμετωπίζουν συνολικά τις πιέσεις, τις προσδοκίες που έχει η κοινωνία από αυτές και ούτω καθεξής. Όντω είναι μεγάλη ισχύ τη δημόσια πολιτική σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Η έκθεσή σας είναι εδώ. Ωραία. Μπορείτε να τη βρείτε λοιπόν και εδώ στο τραπέζι αλλά και στο, στο site μας. Και τώρα Θα μιλήσουμε για τον ιδιωτικό τομέα και την χειραφέτηση των γυναικών στο οικονομικό περιβάλλον. Είναι, θα έρθει η κυρία Γκοζάλους που είναι εκπρόσωπος του ICT. Δεν ξέρω αν θα έχετε αρκετό χρόνο να μας πείτε και να μας εξηγήσετε ακριβώς τι κάνετε. Ίσως θα είναι καλό να ξανάρθετε με τη νέα επιτροπή και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Δερμηνείς που μας έδωσαν ακόμα 10 λεπτά. Δεν θα πάρουμε πάνω από 10 λεπτά. Εάν πάρουμε πάνω από 10 λεπτά, μπορείτε να φύγετε για διάλειμμα. Το λέω από τώρα. Στις 12 και 10 σταματούν οι διερμηνείς να μιλάνε ευχαριστώ. Θα σας αναφέρω σύντομα τις προοπτικές των θεμάτων φύλου από, μια, από ένα άλλο πρακτορείο του ΟΗΕ της υποβοήθησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων διεθνώς, το Διεθνές Εμπορικό Κέντρο. Σήμερα θα σας μιλήσω για τις γυναίκες από οικονομικής απόψεως. Empowerment δηλαδή. Γιατί από οικονομικής απόψεως, διότι 40% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παγκοσμίω ε, αποτελούνται από γυναίκες. Οι γυναίκες 90% των εισοδημάτων τους τα επενδύουν, ενώ μόνο 40 οι άντρες. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η μεγαλύτερη συνεισφορή στην απασχόληση. Από τώρα μέχρι το 2030 θα χρειαστεί να δημιουργηθούν 500 εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης και οι περισσότερες θα είναι από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, αφού μιλάμε για το οικονομικό empowerment των γυναικών, δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, μόνο κοινωνικό θέμα, είναι και οικονομικό. Είμαστε βέβαια οι φυσικοί σας σύμμαχοι για ως προς το θέμα αυτό. Το ΙΕ έχει συντάξει τις κύριες αρχές που διέπουν το θέμα του empowerment των γυναικών. Και θα ήθελα να σας μιλήσω, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα των παρεμβάσεων που κάνουμε και να τελειώσω με τέσσερις συστάσεις που ελπίζουμε πολύ και η Επιτροπή σας να αναλάβει, αν όχι σε αυτή τη θητεία που τελειώνει, τουλάχιστον στην επόμενη. Αρχίζουμε με γυναίκες που καλλιεργούν καφέ στο Βουρούνδι 70% των εξαγωγών του Μπουρούντι είναι καφές και ο περισσότερος από αυτόν τον καφέ καλλιεργείται από γυναίκες. Σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές με λίγες υπηρεσίες και χωρίς πολλή παιδεία για αυτά τα θέματα. Ούτε διασυνδέσεις για τη διάθεση του προϊόντος τους. Τι κάναμε λοιπόν. Θελήσαμε να δούμε ποιες είναι οι δυσκολίες τους και να τους προσφέρουμε λύσεις. Και γι' αυτό συνεργαστήκαμε με τη Διεθνή Συμμαχία Γυναικοκαλλιεργητών Καφέ. Τέτοιες οργανώσεις υπάρχουν στην Τανζανία, στην Ουγγάντα, στον Μπουρούντι, στην Τανζανία για να προωθηθούν αλλαγές στις εφαρμοσόμενες πρακτικές ώστε να μπορέσουν να εμπορευτούν το προϊόν τους διεθνώς. Αναφερθήκαμε σε θέματα συσκευασίας, ποιότητας, ε, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τεράστιο πρόβλημα για τις γυναίκες επιχειρηματίες αυτές και θελήσαμε να διασφαλίσουμε ότι θα διασυνδεθούν επαρκώς με τις διεθνείς αγορές. Αυτά κάνει η οργάνωσή μας. Τώρα τι μαθήματα πήραμε από αυτές τις παρεμβάσεις σε χώρες σαν τον Μπουρούντι με τις γυναικοκαλλιεργήτριες καφέ. Θα μπορούσα να αναφέρω βέβαια και το αμάγκο και τον τουρισμό και το βαμβάκι, αλλά ποια είναι τα τέσσερα μαθήματα που πήραμε από την παρέμβαση αυτή που θα ήταν χρήσιμα και για σας εφόσον συντάσσετε, καταστρώνετε πολιτική στην Ευρώπη. Πρώτον, Οι γυναίκες πρέπει συστηματικά να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις για θέματα που τις αφορούν. Πρέπει να υπάρξουν προγράμματα για γυναίκες με συμμετοχή γυναικών και με ισότητα ώστε να μην διαιωνίζεται το status quo. Παραδείγματος χάρη, όταν βοηθούμε χώρες να εφαρμόσουν αναπτυξιακή, εξωτερική, ε, αναπτυξιακή πολιτική εξαγωγών, λαμβάνουμε υπόψη μας ιδιαίτερα το θέμα των γυναικών. Δεύτερο, έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις επιχειρηματίες. Από τις αναπτυσσόμενες χώρες το έχω δει αυτό, αλλά νομίζω το ίδιο ακριβώς ισχύει και για γυναίκες επιχειρηματίες και στον ανεπτυγμένο κόσμο. Πρόσβαση λοιπόν στη χρηματοδότηση και ιδίως των γυναικών σε τράπεζες. Για τις καλλιεργήτριες καφέ στον Μπουρούντι, οι γυναίκες φυτεύουν και καλλιεργούν τον καφέ, τον πουλούν, αλλά οι άντρες παίρνουν τα εισοδήματα και τα βάζουν στην τράπεζά των. Γιατί διότι οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες. Επομένως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί με μεγάλη προσοχή ώστε οι γυναίκες που όπως σας είπα επενδύουν το 90% των εισοδημάτων τους στην επιχείρησή τους θα έχουν και σωστή διαχείριση των εισοδημάτων τους. Τρίτον, κυβερνητικές προμήθειες. Είναι τεράστιο τμήμα των οικονομιών μας και παρόλα αυτά μόνο 1% των προμηθειών αυτών πηγαίνει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις γυναικών. Αυτό νομίζω δείχνει κάτι και για την Ευρώπη και για αναπτυσσόμενες χώρες και δείχνει ότι πρέπει να αφιερωθούν ειδικά για τις γυναίκες μεγάλα τμήματα προγραμματισμού και πολιτικής. Όπως γίνεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γενικότερα, θέλουμε αυτό να συμπεριλαμβάνει και τις γυναικείες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει βέβαια μερικοί να τα προωθήσουν αυτά και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να γίνει ένας από αυτούς τους υποστηρικτές της υπόθεσης αυτής γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις γυναικών και στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτά τα προγράμματα. Τέταρτον, λογοδοσία και εποπτεία. Ξέρουμε ότι όταν κάτι έχει μετρηθεί εφαρμόζεται. Παραδείγματα μετρήσεων που Κάτι μας πρέπει να προσεχθούν. Η ισότητα των φύλων, η βοήθεια που χορηγείται με βάση την ισότητα των φύλων συγκεντρώνεται σε κοινωνικούς τομείς όπως την υγεία, την παιδεία και πολύ λιγότερο σε οικονομικούς τομείς ή οικονομικές δράσεις οικονομικές. Μόνο το 2% της βοήθειας που χορηγείται στους παραγωγικούς τομείς αφορά την ισότητα των φύλων. Κατ' εμέ λοιπόν μπορούμε να πούμε στην Επιτροπή σας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανάπτυξης, ότι πρέπει να διασφαλιστεί μεγαλύτερο μερίδιο στην αναπτυξιακή βοήθεια Το ΙΤΑ τμήμα του empowerment, το όμικρον γιώτα τμήμα μάλλον, δηλαδή στο οικονομικό empowerment. Ελπίζω, κύριε, Short summary of, um... κύριε Πρόεδρε, ότι με τη συνεργασία όλων των διεθνών αυτών οικονομικών κέντρων θα καταλάβετε ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος διάλογος μεταξύ μας και ζητώ από την Επιτροπή σας να διασφαλίσει ότι μετά το 2015 το αναπτυξιακό πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή συντάσσεται θα βάλει λίγο περισσότερο, περισσότερη έμφαση στο οικονομικό empowerment των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην συνεχιζόμενη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρον θέμα για την επόμενη όμως Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Οι, δουλέ... οι γυναίκες δουλεύουν, αλλά κάποιες φορές ε, αν με λιγότερα χρήματα. Ή άλλοι παίρνουν τα λεφτά τους. και έχετε απόλυτο δίκιο για όλα αυτά που μας είπατε. Θα πρέπει όντως να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Σωστά μας υποδείξατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και πάλι να σας πω ότι λυπούμε που καθυστερήσαμε ναι. αλλά τουλάχιστον τώρα μπορώ να πω ότι κλείνουμε ε, τη συνεδρίασή μας πριν τις 12 και 10. Κλείνουμε την σημερινή συνεδρίαση, είναι τελευταία για αυτή τη θητεία. Θα σας ευχαριστήσω με την ευκαιρία του Σερμινής κατά τη διάρκεια όλης της αιτίας. Ήταν καταπληκτικό ε, που σας είχαμε κοντά μας. Είστε φοβερό εργαλείο και αν θέλετε μπορείτε να βγείτε ε, από τις καμπίνες σας και να έρθετε έξω στο κοκτέιλ ώστε να γνωριστούμε και να συνομιλήσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους.